παραδεισής μου υπάρχει ε, τέλεια σύμπνοια απόψεων ανάμεσα σε εσά και εμένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Κλείνει η συζήτηση για το θέμα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι στις 12. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι προφορικέ ερωτήσεις για την εφαρμογή της στρατηγική τη Ευρωπαϊκής ένωση στην περιοχή του Δούναβη. Έχουμε πέντε συντάκτες που θα λάβουν το λόγο και δίνω το λόγο στην κυρία Τικάου πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη και ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την Ουγγρική Προεδρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Ιανουαρίου του 2010 είχε ψηφίσει ένα ψήφισμα και θα παραμείνει πιστός εταίρος για την υλοποίηση και ενημέρωση της στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή είναι αποτέλεσμα μιας ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τοπικές περιφερειακές αρχές και με εθνικές αρχές, καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με ακαδημαϊκούς κλπ. Και μάλιστα αυτό το τμήμα είναι ακόμη πιο σημαντικό για την υλοποίηση, διότι η στρατηγική αυτή πρέπει να επενδύσει σε καλύτερη πλευσιμότητα, σε καλύτερη διασύνδεση ε, των λιμένων διατροπικών μεταφορών και στην μείωση της ρήπανσης στο Δούναβι. Επίσης θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην αυσιπλοεία, στην εσωτερική αυσιπλοεία η ανάπτυξη τουρισμού και η πρόληψη φυσικών καταστροφών καθώς και η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ε, και της περιβαλλοντικής ρήπανσης θα ε, φέρουν και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στις περιφέρειες αυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή του Ευξήνου Πόντου και πρέπει να έχουμε μια κατάσταση στην οποία όλοι θα βγαίνουν κερδισμένοι όσον αφορά τη βελτίωση της ναυσιπλοείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Χαιρετίζουμε ε, ε, αυτό το οποίο ψήφισαν οι συντονιστές και τους ζητάμε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών και των περιφερειών για να εφαρμοστεί η στρατηγική αυτή το συντομότερο δυνατόν τα κράτη-μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους και να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί προς όφελος αυτής της στρατηγικής. Οι διατάξεις του των ε, ε, πολιετών προγραμμάτων θα πρέπει να λάβουν υπόψη και αυτή την παράμετρο. Μιλάμε για πλωτέ οδού που ενώνουν τη Βόρεια Θάλασσα με την, τον Εύξηνο Πόντο και γι' αυτό θέλουμε η στρατηγική αυτή να επεκταθεί και στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου. Κυρία Μανέσκου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική την περιοχή του Δούναβη είναι μια ενσωματωμένη στρατηγική που θα δημιουργήσει διασυνδέσει μεταξύ των διαφόρων πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιλύσει τα κύρια προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή τη μακροπεριοχή. Η συνεισφορά του η δική μας είναι για να βελτιωθεί η μεταφορά των ε, εμπορευμάτων, η ανάπτυξη των τερματικών σταθμών και τα έργα υποδομής που θα επιτρέψουν στα πολυκομβικά μέσα μεταφορών να βελτιωθούν. Επίσης, θα επιτρέψει να έχουν οι μικρομισές επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια για να μπορέσει η περιοχή αυτή να αναπτυχθεί οικονομικά. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία στην περιοχή ώστε να μπορέσει να υπάρξει αηφόρος ανάπτυξη και να δημιουργηθούν κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δώσει ε, νέες θέσεις απασχόλησης στους κατοίκους της περιοχής, των κρατών μελών εκεί και θα βοηθήσει με εταιρικές ε, σχέσεις ε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση να προβλέψει περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα για να βοηθηθούν όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν στην περιοχή. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς σκέφτεται να εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική η Επιτροπή και ποια είναι η πολιτική την οποία θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σρέντερ, η, η κυρία Σρέντερ, τρία λεπτά, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι μια συνολική στρατηγική για το Δούναβι, για όλες τις περιφέρειες, ε, τους πολίτες και τα κράτη-μέλη είναι ένα τεράστιο όραμα και έχει τεράστια δυναμική για την αηφόρο ανάπτυξη για το σύνολο του ποταμού. Οικονομικές καθώς και περιβαλλοντικές πτυχές θα οδηγήσουν ε, σε αυτό το οποίο θέλουμε τελικά να επιτύχουμε. Η βιολογική και η πολιτιστική πολυμορφία της συνολικής λεκάνης ε, του ποταμού θα μπορέσει να βοηθήσει ε, στην ε, πρόθεση προγραμμάτων και το σημαντικό είναι να φροντίσουμε όλοι να εμποδίσουμε τη ρήπανση του ποταμού. Όλοι θα θυμάστε τις καταστροφές που πολλές φορές έχουν επέλθει σε διάφορες περιοχές του ποταμού. Οι περιοχές ε, και ανάντι και κατάντι του ποταμού θα πρέπει να συνεργαστούν για την κοινή ανάπτυξη του ποταμού διατηρώντας ε, σωστό το περιβάλλον χρειαζόμαστε και την καινοτομία και την πρόοδο επωφελούμενη από τα σφάλματα του παρελθόντος από τα οποία πρέπει να διδαχθούμε και να μην τα επαναλάβουμε και θα πρέπει να προσαρμόσουμε ε, τα σκάφη στον ποταμό και όχι τον ποταμό στα σκάφη. Έχουμε την τεχνική τεχνογνωσία, έχουμε το δυναμικό της περιφέρειας και μπορεί να μας δώσει τεράστιο δυναμισμό και τεράστιες δυνατότητες παγκόσμιας ανάπτυξης από τον ποταμό αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του να διορθώσει την πρόταση της Επιτροπής σε ένα σημείο όπως ε, και στο χώρο της Βαλτικής ε, υπάρχει ένας χώρος διεθνών συμφωνιών ε, για τη συνεργασία σε οδούς εσωτερικές οδούς ναυσιπλοείας και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κοινή δήλωση να έχουμε μια ρήτρα για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και παράλληλα να παραμείνει η δυνατότητα του να είναι πλωτός ο ποταμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και θα πρέπει να το συμπεριλάβει η Επιτροπή. Για να το επιτύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και οπωσδήποτε διαφάνεια το έχουμε δει από την εμπειρία μας μέχρι τώρα ότι η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά ούτω ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον ποταμό για τις επόμενες γενιές, για αυτούς οι οποίοι ζουν και εργάζονται κατά μήκος του ποταμού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια για να μπορέσουν να προωθηθούν τα μέτρα αυτά. Τα σφάλματα του παρελθόντος θα πρέπει τώρα να τα διορθώσουμε και να έχουμε μια ισορροπημένη συνεργασία και οικονομική και περιβαλλοντική για όλη τη λεκάνη του ποταμού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Βλασάκ. Κύριε Επίτροπε, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι πρώτα απ' όλα ένα πολιτικό εργαλείο είναι μία από τις ε, πιθανές μορφές συνεργασίας και θα πρέπει να οδηγούν σε καλύτερη χρήση των ε, πρωτοβουλειών, των ε, προγραμμάτων, των πλατφορμών συνεργασίας. Οι μακροπερφιακές στρατηγικές θα πρέπει επίσης να αποτελούν ένα πλαίσιο για την καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς και μία πλατφόρμα για τη δημιουργία επιχειρηματικών συνδέσμων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων θα πρέπει να οδηγούν σε εξυγχρονισμό και σε καλύτερη ε, διάρθρωση, σε καλύτερες διαρθρώσεις, ούτως ώστε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Τα μέσα αυτά όμως, τα μακροπεριφερειακά, θα πρέπει να ορίζονται καλύτερα. Ε, γι' αυτό η έννοια των μακροπεριφερειακών στρατηγικών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν συστηματικό τρόπο ούτως ώστε να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση για το θέμα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αριθμό των στρατηγικών, τη συγκέντρωσή τους, τον χαρακτήρα τους και την ε, ε, διοίκησή τους. Η έννοια ε, παρομοίων στρατηγικών, μεταξύ των οποίων και ε, η υποσυζήτηση μας βρίσκει σύμφωνους αν βασίζεται στις βασικές αρχές της δημοσιονομικής και νομοθετικής ουδετερότητας και της θεσμικής ουδετερότητας. Ο ρόλος και το μέλλον των μακροπεριφερειακών στρατηγικών σχετίζεται στενά με τη συζήτηση για τον, τη μελλοντική χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων. Σίγουρα όμως υπάρχει μια επικάλυψη και με την συζήτηση για το μέλλον των θεσμικών μας πολιτικών. Δεν θα πρέπει να προδικάζουμε ε, το αποτέλεσμα των ε, μελλοντικών, ε, των επόμενων ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Γι' αυτό ανησυχώ κάπως οι μακροπεριφερειακές αυτές στρατηγικές δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την μελλοντική δομή των πολιτικών συνοχής ή τον καταμερισμό των κονδυλίων στους επιμέρους στόχους μας. Ο κύριος Ντόιτς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πράγμα συζητάμε όταν μιλάμε για την ε, περιφέρεια του Δούναβη. Η περιφέρεια του Δούναβη καλύπτει 14 ε, χώρες ε, και 160 πολίτες της Ευρώπης και ενώνει χώρες και πολίτες. πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η στρατηγική της Ευρώπης για το Δούναβι είναι μια στρατηγική του μέλλοντος. Και είναι η στρατηγική όχι μόνο για την κεντρική Ευρώπη, αλλά μια στρατηγική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια στρατηγική που κατευθύνεται στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Κατά τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Περιφέρεια του Δούναβη χρησιμοποίησαμε μια παλαιά μέθοδο. Μπορούμε σιγά σιγά να φέρουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στους πολίτες. Και γι' αυτό τώρα έχουμε οργανώσει διαβούλευση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι προέκυψε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η στρατηγική αυτή είναι πολύ σημαντική για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες κατά μήκο του Δούναβη έχουν πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση και γι' αυτό η στρατηγική για το Δούναβη θα πρέπει να είναι μια στρατηγική που θα αντισταθμίζει τις απώλειες από την οικονομική κρίση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να χαιρετήσουμε τις προσπάθειες της Ουγγρικής κυβέρνησης για την ε, προσέγγιση ε, των ε, πολιτών και θα πρέπει να προωθήσουμε τη συνεργασία όλων ούτως ώστε όλες οι εμπλεκόμενες χώρες να επωφεληθούν και από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή τι έχει να μας πει για την στρατηγική του Δούναβη, ο Επιτροπός κ. Χάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή με μεγάλη χαρά ασχολήθηκε με αυτό το θέμα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αφορούν ε, τις εμπλεκόμενες χώρες και τις περιοχές αυτές και έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική όπου ε, θελήσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών ε, μελών ε, και να βελτιώσουμε το επίπεδο διαβίωσης όλων. Ε, μιλάμε για κινητικότητα, βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων και μέσω αυτών και ενίσχυση της ευημερία. Αυτή είναι μια νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη στρατηγική μας. Είναι ε, σημαντικό ότι έχουμε συμπεριλάβει την ενεργό συμμετοχή όλων ε, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και την κοινωνία των πολιτών και την οικονομία διότι θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν και ο χώρος του Δούναβη φαίνεται ότι είναι ο κατάλληλος χώρος για τη συνεργασία αυτή. Χρειαζόμαστε αηφόρο ανάπτυξη και γι' αυτό έχουμε από τους 11 τομείς προτεραιότητες τρεις που ασχολούνται με την βελτίωση της ποιότητας του ύδατος και με την προστασία της φύσης ε, και εδώ συμπεριλαμβάνονται και η πρόληψη των πλημμυρών που θα πρέπει να φροντίσουμε σε όλο το μήκος του Δούναβη είναι ο πλέον διεθνής ποταμός σε ολόκληρο τον κόσμο ο Δούναβης. Δέκα χώρες ε, βρίσκονται κατά μήκο του Δούναβη. Κανένα άλλο ποταμό σε ολόκληρο τον κόσμο δεν έχει τόσες πολλές χώρες κατά μήκο του. Είναι σημαντικό και θα πρέπει να υποφεληθούμε από την ευκαιρία αυτή όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, μια, μακρο, μακροοικονομική στρατηγική ε, μεταξύ των χωρών που βρίσκονται κατά μήκος του Δούναβη είναι ε, οκτώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέσα τα οποία διατίθεται θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καταλήλως για να επωφελήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Θα πρέπει με έξυπνο τρόπο να συνδυάσουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα με το στόχο να προωθήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα στις διάφορες ε, περιφέρειες. Σε πολλές ε, συζητήσεις ε, και πολυμερείς και διμερείς το τονίζουμε αυτό και τώρα που προετοιμάζουμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το είδος των προγραμμάτων τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε σε σχέση συνεργασίας και τους πόρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει τα μέσα τα οποία διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 30 ε, εκατομμύρια ευρώ, ε, ε, ευρώ να, να τα χρησιμοποιήσουμε. Από πλευρά της Επιτροπής θα υποστηρίξουμε αυτή την πολιτική και υπάρχει μια ομάδα υψηλού επίπεδου στην οποία ε, τακτικά υποβάλλεται έκθεση και παρακολουθούνται τα θέματα αυτά με συσκέψεις και με εκθέσεις ούτως ώστε να δοθεί μια συνολική υποστήριξη σε όλα αυτά τα θέματα και προσπαθούμε να ε, συμπεριλάβουμε σε αυτήν την προσπάθεια όλους αυτούς που βρίσκονται επί τόπου ούτως ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να μπορέσουν να εφαρμοστούν σωστά και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα έχουμε τις παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Μαρινέσκου για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εκ μέρους του ΕΛ θα ήθελα να πω ότι με ευχαρίστηση λάβαμε υπόψη το έγγραφο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγκριθεί για τη διάρκεια της παρούσης Προεδρίας. Είναι για να μπορέσει να αναπτυχθεί η στρατηγική στην περιοχή να κάνουμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να έχουμε κατάλογο πρωτοαιρετήτων. δεύτερον συντονισμό όλων των δράσεων της Κομισιόν και τρίτον πόρους για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα προγράμματα και οι δράσεις. Είπα ότι θα πρέπει να έχουμε με ένα κοινό κατάλογο σχεδίων εκ μέρους όλων των ε, παραδουνάβιων κρατών. Αυτό για να μπορέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο να συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και να κάνουμε την περιοχή πιο ελκυστική. Γι' αυτό θα πρέπει το σχέδιο αυτό με τις κοινέ στρατηγικές συγχρόνως να τις εφαρμόσουμε παντού. Πιστεύω ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στρατηγική της στρατηγικής Βαλτικής απέδειξε ότι για να αποδώσει θα πρέπει να υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει τα συμπεμφωνημένα να υλοποιηθούν. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση και μία στρατηγική βάση κοινού καταλόγου προτεραιοτήτων και συντονισμένες προσπάθειες. Υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται, υπάρχουν τα ε, διαρθρωτικά σχέδια, αλλά θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να μπορέσουμε επίσης και να μεταφέρουμε μη χρησιμοποιημένα κονδύλια για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ταμπάντζη εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο Επίτροπος κ. Χάν ε, προέρχεται από μια χώρα που βρίσκεται κατά μήκο ε, του Δούναδη. Και παράλληλα υπάρχει και η Ουγγρική Προεδρία που επίσης ε, αποδίδει σημασία σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες, αγαπητοί συνάδελφοι. Και δεν είναι εύκολο να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Δεν το λέω γιατί έχω αμφιβολίες και βέβαια θέλω να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Και το θετικό στη στρατηγική αυτή είναι ότι υποχρεώνει τις παράκτιες, ε, τις παραποτάμιες χώρες να συνεργαστούν στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Οι στόχοι μας συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα του ύδατος, ε, την δυνατότητα πλεύσης ε, του ποταμού, την προστασία του περιβάλλοντος, τον οικοτουρισμό, είναι προτεραιότητες τις οποίες ε, μπορούμε να έχουμε εξισορρόπηση όλων των παραμέτρων ώστε να επιτύχουμε κάτι το επωφελές για όλους. Η κυρία Χαουσμένοβα, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη πρόκειται να εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών τον ερχόμενο Απρίλιο και αυτό θα αποτελέσει ένα μήνυμα προς την κοινή γνώμη ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια για την εφαρμογή της. Στην πράξη όμως, ε, κράτη μέλη και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια στο συντονισμό των προτεραιοτήτων και των μηχανισμών για την εφαρμογή και τον έλεγχο αυτής της στρατηγικής. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μεγάλα διασυνοριακά έργα και προγράμματα. Ε, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην παρακολούθηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ε, στην τήρηση των προθεσμιών και στην ε, ε, επίδευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι ευθύνε και οι αρμοδιότητε θα πρέπει να καθοριστούν σαφώ, η υποβολή εκθέσεων και οι αναλύσει επίση. Ένα άλλο βασικό πρόβλημα είναι η επικοινωνία και η δημοσιοποίηση ε, των αποτελεσμάτων και βεβαίω η εφαρμογή τη στρατηγική. Η διαφάνεια και η πρόσβαση στην ενημέρωση είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντε, καθώ επίση και οι εσωτερικέ διαδικασίες μεταξύ των συντονιστών. Πριν από την ε, στρατηγική αυτή έγιναν ε, εκτεταμένες συζητήσεις όσον αφορά τις προτεραιότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η στρατηγική. Αυτό προκάλεσε αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως οι πολίτες πώς θα ενημερωθούν για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Αυτό είναι ένα ερώτημα που περιμένει την απάντησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ευαισθητοποίηση πρέπει να ε, συνεχιστεί μέσω ειδικών εκστρατιών μέρος της κοινή γνώμης. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόχ Μπίλερ, μέρος των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό η επεξεργασία αυτής της στρατηγικής να είναι μια ανοιχτή διαδικασία δεν θα πρέπει μόνο λίγοι φορείς ε, να παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να συνδυάσουμε ε, αντιτιθέμενα ενδιαφέροντα. Θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας το συνδυασμό των οδικών με τις πλωτές μεταφορές και να βρούμε τις σωστές λύσεις για την περιοχή του Δούναβη. Να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές δυνατότητες για να προσαρμόσουμε τα σκάφη στον ποταμό και όχι το αντίστροφο εδώ έχουμε μια ανακοίνωση της Επιτροπής που θα πρέπει να ε, λαμβάνει υπόψη ε, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να υποστηρίξει αυτά τα οποία υπάρχουν. Η ε, Επιτροπή μιλάει για σκάφη της κατηγορίας 4β τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να πλέουν πράγμα το οποίο αποτελεί κάτι που δεν είναι συμβατό με τις υφιστάμενες τεχνικές ε, δυνατότητες. Αυτό είναι μια διάταξη που θα πρέπει να αποσυρθεί και επιπλέον θα ήθελα να τονίσουμε ότι η στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά θα πρέπει να τη συνδυάσουμε με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ε, ανακοίνωσή της και το σχέδιο δράσης για το Δούναβι και το τμήμα 2.1 μιλάει για τη στρατηγική και για τις ευκαιρίες και για το πώς αυτές οι χώρες μπορούν να συνεισφέρουν για την ανάπτυξη αυτής της περιφέρειας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη του Δούναβι για τις αποτελεσματικές ε, μεταφορές. Κατανοούμε ότι η δυνατότητα δυνατότητα εκμετάλλευσης του ποταμού για αυτούς τους σκοπούς ε, δεν, ε, έχει εκμεταλλευτεί, δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρων από το Βλαντιβοστόκ μέχρι τη Βιέννη ή την Πρατισλάβα. Θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό ε, να εφαρμοστεί σωστά για να βελτιώσει την πλευσιμότητα του Δούναβη. Είναι πολύ σημαντικό και θα δώσει μια τόνωση τη οικονομία και τη ανάπτυξη στην περιοχή. Πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε για να μπορέσουμε ε, να λάβουμε υπόψη μα και του κινδύνου πλημμύρα και να βελτιώσουμε τι δυνατότητε που υπάρχουν, να βελτιώσουμε την πλευσιμότητα του ποταμού και να δημιουργήσουμε επίση ενέργεια από ανανεώσιμε πηγές. Είναι προγράμματα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από διάφορους πόρου και από το Ταμείο Συνοχής εφόσον βρούμε το σωστό μηχανισμό για να γίνει δυνατό κάτι τέτοιο. Ο κύριος Βανίστερ Ρόι. Κύριε ε, ε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Είναι θετική η πρόταση για την περιοχή του Δούναβη. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ε, που είναι η διάβρωση των εδαφών και ένα ακόμα πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν ε, αξιοποιούμε πλήρως την ε, δυναμικότητα αυτής της περιοχής προς όφελος των πολιτών μας. Ως Ολλανδός γνωρίζω ότι έχουμε υιοθετήσει μια σχετική προσέγγιση για το Ρήνο και ότι αυτό είχε θετικές συνέπειες, θετικές επιπτώσεις και για την γεωργία και για τον τουρισμό. Τώρα, Ποια είναι η βάση για την ε, βελτίωση της εδαφικής συνοχής. Αυτό περιλαμβάνεται μέσα στη συνθήκη και αυτό το νέο άρθρο επιτρέπει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 14 χωρών. Υπάρχει ο στόχος 3 της πολιτικής συνοχής που αποτελεί μια εξαιρετική βάση και ε, οι τοπικές κοινωνίες, οι πολίτες θα, μπορέσουν έτσι να εμπλακούν. Το ΕΛ λέει ναι στις τρεις αυτές προϋποθέσεις, όχι νέες δομές, όχι νέο νομοθετικό πλαίσιο, όχι ξεχωριστό ταμείο, όπως το υπενθύμησε και ο Επίτροπος. Αξιοποίηση διαθέσιμων ε, ταμείων και κονδυλίων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων οι μακροπεριφέρειες δεν πρέπει να γίνουν πιο πολύπλοκες. Η βάση πρέπει να είναι η περιφέρεια, τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τα υπάρχοντα μέσα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εργαστούμε αποτελεσματικά με ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης. Το Συμβούλιο ε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ξεκίνησε ήδη μια τέτοια στρατηγική για την Βαλτική θάλασσα. Τώρα έχουμε το Δούναβι. Ε, ακολουθεί ο Ατλαντικός. Ε, συναντήθηκα σήμερα το πρωί με φοπλιστές Ολλανδούς οι οποίοι μου είπαν ότι αν γίνει διεύρυνση των, και επέκταση των πλωτών οδών ε, θα μπορέσουμε να έχουμε 10% μεγαλύτερη ανάπτυξη ε, αν αξιοποιήσουμε περισσότερο τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα. Ευχαριστώ. Into a continuing process and into a tool for coordination among partners. Ο κύριος ε, Κυρίλο, ε, θα πρέπει να βελτιωθεί στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ε, η εφαρμογή κοινών στόχων και θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση οι πολίτες μας για μια τόσο μεγάλη, ε, μεγάλη σημασία ευρωπαϊκή στρατηγική. Ε, επίσης, ε, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω και θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός με την πολιτική συνοχής. Η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων είναι η εγγύηση ότι όλοι θα αναγνωρίσουν σε δικιά τους προτεραιότητα τα προγράμματα δράσης και τις στρατηγικές αυτές οι περιφέρειες ε, ε, του Δούναβη ε, θα πρέπει να δώσουν χρήματα από το δικό τους προϋπολογισμό. Αυτό θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να γίνει ένα καλό παράδειγμα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σερνάλοβα έχει το λόγο. και προέρχεται από μία από τις ε, περιοχές ε, ε, των παραπόταμων του Δούναβη. Ναι, όντως, κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική του Δούναβη αποτελεί άλλη μία μακροστρατηγική, μακροπεριφερειακή στρατηγική που θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα σωστή συνεργασίας μεταξύ χωρών που έχουν κοινά συμφέροντα. Συμφωνούμε ότι ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η αηφόρος ανάπτυξη χρησιμοποιώντας τα μέσα και τις πολιτικές που έχουμε στη διάθεσή μας. Όχι στη γραφειοκρατία, όχι σε νέους θεσμούς και όχι σε θεσμικά κονδύλια. Τρία όχι λοιπόν. Αλλά παράλληλα έχουμε και μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Πώς θα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σωστή εφαρμογή αυτής της στρατηγικής στην πράξη Ιδίω σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και με τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η επικουρικότητα και θα πρέπει να συνδυάζονται όλα αυτά τα επίπεδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνδυάζει αυτές τις προσπάθειες και η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την υλοποίηση. Η ερώτησή μου είναι αν θα υποβάλει η Επιτροπή μια πιο πλουστευμένη, πιο ευανάγνωστη μορφή αυτού του κειμένου που να βοηθά τους ανθρώπους επιτόπου. Και άλλη μια ερώτηση, πώς θα συνδεθεί με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών προοπτικών μέχρι το 2020 αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ κυρία Κάντενμπαχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Υπάρχουν 11 τομείς προτεραιότητες ε, και ε, μας χαροποιούν όλα αυτά. Η στρατηγική για το Δούναβι είναι μια στρατηγική που ξεκινά από τη βάση προς τα πάνω και αυτό εξαρτάται και από τις χώρες της παραποτάμιας και από τους πολίτες που όλοι θεωρούν σημαντική αυτή τη στρατηγική για το Δούναβι. Παρακολουθώντας τη συζήτηση σήμερα φαίνεται σαφώς που βρίσκονται οι μεγαλύτερες ανησυχίες. Νομίζω ότι θα Πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά ε, την πολιτιστική συνεργασία. Σωστή συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα πάντοτε υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει. Πρόβλημα υπάρχει στην βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Πολύ συχνά βλέπουμε το Δούναβι ως ε, πλωτή οδό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να βλέπουμε και τους κινδύνους για το ε, περιβάλλον και να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος ή τουλάχιστον αυτό είναι πολύ φιλόδοξο να μην αυξηθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Θα πρέπει να σκεφτούμε ε, και ε, όλο το οικοσύστημα το οποίο βρίσκεται γύρω από το Δούναβι και ε, στους παραποτάμους του και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό απαιτεί και αρκετούς οικονομικούς πόρους αλλά είναι πια θέμα του, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να μπορέσουν τα μέσα τα οποία είναι αφιερωμένα στο Δούναβι να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά ούτως ώστε και ο Δούναβης και οι παραπόταμοι του ε, και οι υδροβιότοποι να είναι τμήμα μια μεγάλη πολιτική αηφόρου ανάπτυξη. Αυτό είναι μια πρόκληση αν θέλουμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη. Γιατί η στρατηγική για το Δούναβι μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε πραγματικά σε πράσινε τεχνολογίε, μα δίνει τη δυνατότητα να τοίσουμε την αηφόρου ανάπτυξη από τη βάση προ τα πάνω. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα δώσει αυτό το οποίο περιμένουν οι πολίτες επιτόπου και όλοι θα πρέπει να, χρηματο... να χρησιμοποιήσουμε τι δυνατότητε και να δώσουμε το παράδειγμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουν όλοι. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κάντενβαχ. Κύριε Σκάλφιν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, από την αρχή ε, η στρατηγική αυτή για το Δούναβι θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα για τις χώρες του Δούναβι. Ε, υπάρχουν πολλές ιδέες στις χώρες ε, γύρω από το Δούναβι, αλλά οι αρχικές προτεραιότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κοινή τουριστική κοινέ τουριστικέ ε, διαδρομέ, ανάπτυξη των ε, μεταφορών. Πρέπει να έχουμε εκεί ορατά αποτελέσματα. Πρέπει να τονίσω ακόμη μια φορά την ανάγκη συμμετοχή των δομών τη Κοινωνία των πολιτών από την πρώτη αρχή. Η στρατηγική αυτή θα επιτύχει όταν οι πολίτε ε, κατά μήκο του Δούναβη θα συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων μορφών συνεργασία που του προσφέρονται. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση και προς την Κομισιόν και προς τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανοίξουμε γραφεία ε, ενημέρωσης, να συνεργαστούμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πανεπιστήμια για να έχουμε ε, χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχουμε χρόνο ε, μόνο για πέντε ομιλητές και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια επιλογή. ο κύριος Μικολάση έχει πρώτα απ' όλα το λόγο by mohla byť... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ευχαριστώ. Η στρατηγική για το Δούναβι θα είναι κενό γράμμα αν δεν την εφαρμόσουμε με το σωστό τρόπο. Και ακριβώ αυτό συζητάμε απόψε. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι είναι θετικό ένα τέτοιο πρόγραμμα διατροπικών ε, μεταφορών ε, να αποτελεί τμήμα αυτή τη στρατηγική. Το λιμάνι τη Μπρατισλάβα θα είναι σημαντικό τμήμα αυτή τη όλη στρατηγική ούτως ώστε να μην αποδίδουμε μεγάλη σημασία ε, να μην έχουν μεγάλο ρόλο οι οδικέ μεταφορέ, δεδομένη τη μεγαλύτερη ρήπανση που προαρχείται από τι οδικέ μεταφορέ. Με τη συμμετοχή του πρώην ε, Επιτρόπου κ. Φιγκέλ σε μια διάσκεψη που έγινε, τονίσαμε τη σημασία τη όλη αυτή τη περιφέρεια και τη συμμετοχή στη στρατηγική για το Δούναβι. Τα θέματα του περιβάλλοντος και της πρόληψης των φυσικών καταστροφών είναι βασικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή δεν θα έχει επιπτώσεις ε, όσον αφορά τα μέσα τα οποία διατίθενται από τα διορθωτικά ταμεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε μετά από το 2004 και το 2007 για την περιοχή του Δούναβη σαν μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υιοθέτησε μια ειδική στρατηγική η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Δούναβη. Ξέρουμε βεβαίως ότι θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν για να ευνοηθεί η περιοχή μέσα να αναπτυχθεί και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Είναι πρωταρχική σημασίας οι διάφορες διαφορές μεταξύ των χωρών των παραδουναβίων να ξεπεραστούν και να δοθούν τα απαραίτητα κοινοτικά κονδύλια. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα το ενεργειακό. Ο κατακαιρματισμός της ενεργειακής αγοράς είναι κάτι το οποίο αυξάνει το κόστος και δεν οδηγεί σε υγιή ανταγωνισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσει να υπάρξει μία ενιαία εσωτερική αγορά που να εγγυάται την ενεργειακή ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Κύριε Σαμπεμάιερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση του δικτύου μεταφορών και των ε, ε, υποδομών καθώς και βελτίωση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό χρειάζονται σωστά προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιούν τη σωστή περιβαλλοντική τεχνολογία. Αυτό το οποίο όμως δεν υπάρχει είναι το θέμα της ασφάλειας για το περιβάλλον σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Ένα ένας από τους σταθμούς στο Βασόμιλε Πεσίστη βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή αυτή του Δούναβη και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και παρότι οι συνέπειες είναι διασυνοριακές από αυτό το σταθμό πυρηνικής ενέργειας δεν λαμβάνονται ε, υπόψη οι διαμαρτυρίε των γειτονικών περιοχών και δεν ε, έχουν επαρκώ ληφθεί υπόψη στην όλη διαδικασία διαβούλευση. Υπάρχουν περιβαλλοντικές τάσεις μεταξύ γειτονικών ε, χωρών και περιφερειών και θα έπρεπε μέσω αυτής της στρατηγικής να αρθούν αυτές οι δυσκολίες που υπάρχουν. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Μεσάρος. Ευχαριστώ.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 Ε, όταν ε, ήμουν παιδί και πηγαίναμε ε, στο Δούναβι για μπάνιο, πολύ συχνά χτυπούσα τα γόνατά μου και τραυματιζόμουν. Ελπίζω να μην υπάρχει πλέον ο κίνδυνος από, το Δούναβι για, για τους λουόμενους και για τους πολίτες που ζουν γύρω από το Δούναβι, βελτιώνοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ποιότητα των υδάτων. Πιστεύω ότι είναι κρίμα που δεν μπορούν να δοθούν επιπλέον μέσα και πόροι. Οι διαφορές είναι μεγάλες μεταξύ των παράκτιων των παραποτάμιων χωρών και είναι σημαντικό να δούμε ότι ο Δούναβης ενώνει παλαιά και νέα κράτη-μέλη. Και Μέσω της στρατηγικής για το Δούναβι μπορούμε να βελτιώσουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις εμπειρίες μας και ε, για τον έξινο πόντο μπορούμε να επωφεληθούμε. Κυρία Ντανσέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Δούναβη βάσει της ε, στρατηγικής της Βαλτικής και με συντονισμό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς είναι πολύ θετική διότι θα επιτρέψει στη περιοχή αυτή να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της επιδοχής. Οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών ε, της περιοχής θα μειωθούν. Οι συνθήκες ε, πλευσιμότητας του δούνομι θα βελτιωθούν. Θα δημιουργηθεί ένας, ε, μια διαρκής πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των περιοχών και μακροπρόθεσμα θα υπάρξει ε, όφελος περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό. Θέλουμε να υπάρξουν νέε επενδύσει για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά αυτή η νέα στρατηγική που θα βελτιώσει το επίπεδο και την ποιότητα ζωή όλων των πολιτών τη Ευρώπη που ζουν στι παραδουνάβιε περιοχέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έφτασε τώρα η ώρα να απαντήσει ο Επίτροπος κ. Χάν στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις σας. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχω λίγο χρόνο δεν θα μπορέσω να απαντήσω στα πάντα, θα ήθελα όμως σε μερικά πράγματα να απαντήσω. Το θέμα της πλευσιμότητας ε, του ποταμού είναι ένα σημαντικό θέμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, όλες τις ε, οικολογικές και οικονομικές παραμέτρους ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, να συνδυάσουμε έξυπνα όλες τις πτυχές και να μπορέσουμε να λάβουμε τα σωστά τεχνολογικά μέτρα, ώστε να έχουμε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη επιβάρυνση της κήτης του ποταμού και επίσης πρέπει να πω ότι εγώ είμαι από ε, είμαι από αυτούς που συμφωνούν ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα σκάφη στον ποταμό και όχι τον ποταμό στα σκάφη είναι σαφές ότι δεν πλέουν τα ίδια σκάφη στο Δούναβι, στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη ε, τα θέματα και αποστάσεων των μεταφορών. Μιλάμε για αποστάσεις γύρω στα 100 χιλιόμετρα και είναι ενδιαφέρον ε, να δούμε και το μέγεθος των σκαφών για να δούμε ε, αν μπορούμε να εφαρμόσουμε ή να προσφέρουμε τα σωστά μεγέθη σκαφών ανάλογα και με την απόσταση που διαπλέουν συνήθως στις διάφορες περιοχές. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης ε, όσον αφορά ε, τη μακροπεριφέρεια του Δούναβη και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και θα πρέπει και όλα τα τμήματα της κοινωνίας των πολιτών να συμπεριληφθούν ενεργά στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και συμφωνώ με αυτά που είπε και η κυρία Κάντενμπαχ και άλλοι βουλευτές ε, ότι ε, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για τη στρατηγική αυτή. Αυτόν τον ενθουσιασμό θα πρέπει να τον ε, διοχετεύσουμε κατά το σωστό τρόπο ούτω ώστε και οι πολίτες να συμμετάσχουν και θα πρέπει να εφαρμόσουμε τώρα τα μέσα τα οποία θα υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τις οποίες έχουμε δώσει. Και γι' αυτό κάνω έκκληση προς όλους ώστε να υλοποιήσουμε σωστά τις πολιτικές αυτές. Υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι και τους, τους διαθέσιμους πόρους θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε σωστά και έξυπνα για να αποκομίσουμε τη σωστή προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουμε τους πολίτες, τα 160 εκατομμύρια πολιτών που ζουν κατά μήκος του Δούναβη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Κλείνει η συζήτηση το θέμα αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει την 5η το μεσημέρι στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής